Colleagues, please be seated. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε παρακαλώ στις θέσεις σας. Okay, thank you. Good morning. Καλημέρα σας λοιπόν και ευχαριστώ. Μετά από ένα διευρυμένο προεδρείο που κράτησε αρκετή ώρα και δεν έχει ακόμα τελειώσει, θα συνεχιστεί αναγκαστικά με τη γραπτή διαδικασία, θα ήθελα να κήρυξουμε την έναρξη της τακτικής μας συνεδρίασης. Καλωσορίζω τους συναδέλφους, τους προσκεκλημένους. Με τα συνέχεια διαδικαστικά ξεκινώ. Υπενθυμίζω ότι έχουμε διαδικτυακή μετάδοση της συνεδρίασης. Ως προς την ε, διερμηνία, προτεραιότητα δίδεται στις γλώσσες των τακτικών μελών της Επιτροπής μας. Η μερίσια διάταξη, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνεται και πρακτικά. Έχετε λάβει τα πρακτικά προηγουμένων συνεδριάσεών μας και συγκεκριμένα ε, της 3ης και 4ης Μαΐου του 2017 και της ε, 8ης Ιουνίου. Μέχρι το τέλος της συνεδρίας έχετε περιθώριο να καταθέσετε σχόλια, παρατηρήσει διορθώσεις. Εάν δεν κατατεθούν σχόλια, παρατηρήσει διορθώσει, θεωρούμε ότι εγκρίθηκαν και τα πρακτικά και σας ευχαριστώ. Και τώρα θα περάσω σε ένα σημείο που αφορά την επίσκεψή μου στο Κίεβο και την Ανατολική Ουκρανία για να σας ενημερώσω. από τρεις πολιτικές ε, ομάδες, η ο κύριος Όστρεβίτσιος εκ μέρου της ε, Άλντε, η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς εκ μέρου των Πρασίνων, η οποία κυρία Χάρμς έλαβε μέρος και στη συνεδρίαση, έλαβε μέρος στη συνεδρίαση στο Κίεβο, ε, ενώ υποφαινόμενο και ο κύριος Οστρεβίτσιος ήμασταν και ήμασταν στην Ανατολική Ουκρανία. Πήγαμε με το τρένο στο Σλόβενσκ, μετά πήγαμε στο Μάγιορσκ. Και κάναμε και τα 700 χιλιόμετρα των κατεχομένων για να φτάσουμε στα κατεχόμενα μέσα σε μία μέρα. με ιδιαίτερες δυσκολίες στην ε, Αφνιέφκα, μετά στον Δνήπερο κοντά ήταν η διανυκτέρευση, επιστρέψαμε μετά στο Κίεβο. Ε, είχαμε συνάντηση με την Μετσλίστη Διεθνές Συνέλευση των Τατάρων της Ουκρανίας. της Κρυμαίας, συγγνώμη. Και βέβαια διαπιστώσαμε μια κατάσταση δύσκολη. Συναντηθήκαμε με τον Μουσταφά Τζεμιλεύ, ο οποίος μας ενημέρωσε για την κατάσταση στην Ουκρανία. Το εφάτου Τσουπάρεφ, ηγετική μορφή επίσης, που έχουμε επανειλημμένα συναντήσει στις αποστολές μας. και συμφωνώ με τις προτάσεις του Μάικλ Μίχαελ Γκάλερ, ότι θα χρειαστεί οπωσδήποτε ένα τέτοιο ταξίδι να το επαναλάβουμε. Αυτά. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω παραπάνω. Θέλω μόνο, αν μου επιτρέπετε, να περάσω στο πρώτο θέμα της ουσίας της συζήτησής μας που αφορά ανταλλαγή απόψεων. σχετικά με την προστασία των διαστημικών αποδομών για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν καλωσορίζω τους τρεις διακεκριμένους ομιλητές μας τον κύριο Αλέν πρώτο, Γενικό Διευθυντή της ε, EU του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκμετάλλευση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων, που ασχολούνται με τη μετεωρολογία και την πρόβλεψη του καιρού. Μετά τον γνωστό σε όλους σας Φιλίπ Μπρουνέ, διευθυντή της Γενική Διεύθυνση Grow και εν τέλει, ιδιαίτερος καλωσορίζω, τον κύριο Ρόλφ Τένσιν, διευθυντή επιχειρήσεων και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαστημικών Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Επιτρέψτε μου λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Αλενατία, τον πρώτο μας ομιλητή. Παρακαλώ. Thank you very much for giving... Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Θα σας δώσω την οπτική γωνία ενός φορέα δορυφόρων. Θα σας παρουσιάσω πρώτα απ' όλα τι είναι η EUMETSAT, ώστε να καταλάβετε για ποιο λόγο είναι ζωτική σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες και η υποδομή. Είμαστε ένας διακυβερνητικό οργανισμός με 30 κράτη-μέλη, δηλαδή έχουμε κράτη-μέλη και πέραν τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία, Ισλανδία. Επόμενη διαφάνεια, έχουμε 9 δορυφόρου σε τρόχια αυτή τη στιγμή. Αποστολή μας ε, συνοπτικά είναι η παρατήρηση και υποστηρίζουμε την πρόβλεψη του καιρού αλλά και την ποιότητα του αέρα και των ωκεανών και την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε τις δικές μας αποστολές, 9 δορυφόρους ε, τροχιά, 6 είναι ιδιόκτητοι για τον καιρό κυρίως, ε, αλλά κάνουμε και αποστολές ε, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Κοπέρνικος. Η υποδομή αυτή είναι ζωτική σημασία για του Ευρωπαίου πολίτε, όπω θα δείτε, διότι παρακολουθούμε ε, σε πραγματικό χρόνο τον καιρό και ειδικότερα ε, καιρικέ συνθήκε που απειλούν την ασφάλεια ε, ή την ιδιοκτησία, των πολιτών. Εδώ βλέπετε τον καιρό σε πραγματικό χρόνο, όπως βλέπετε. Εδώ βλέπετε μια καταιγίδα στην Ευρώπη. Θα μπορούσα να σας δείξω και κάποια αμοθίελα, για παράδειγμα στο Αφγανιστάν ή αλλού, ε, ε, φαινόμενα που επηρεάζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και που παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό. Ένα άλλο παράδειγμα εδώ, όχι πάμε πίσω. Εδώ βλέπετε στάχτη, ε, ένα σύννεφο στάχτης από ηφαίστεια πολύ σημαντικό για τη διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας. Εδώ βλέπετε γεωστατική τροχιά, ε, τον καιρό δηλαδή σε πραγματικό χρόνο και εδώ βλέπετε και ένα ε, σύστημα ε, τροχιάς, το Polar System που το λειτουργούμε μαζί με τη ΣΥΠΑ. Εμείς λειτουργούμε σε μια τροχιά και συμπληρωματικά η ΕΠΑ λειτουργούν σε μια άλλη τροχιά και ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Είναι ένα πραγματικά ολοκληρωμένο σύστημα διπλής χρήσης. Ε, η δορυφόρη αυτή είναι πολύ σημαντική για οποιαδήποτε πρόβλεψη έως και 12 ημερών. Και χάρη στους δορυφόρους αυτούς είναι δυνατή η πρόβλεψη ε, ίδιας ποιότητας ε, οπουδήποτε στον κόσμο καθημερινά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις διάφορες επιχειρήσεις. Κάποια ζητήματα πολιτικής, ε, κάποια στοιχεία πολιτικής. Αυτό είναι σημαντικό διότι ε, εδώ έχουμε τη γεωσκόπηση και την παρακολούθηση του καιρού που έχουν κάποια κοινά ζητήματα. Όταν παρακολουθεί κανεί τον καιρό δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Καμία χώρα δεν μπορεί να κάνει τα πάντα μόνη τη. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα παγκόσμιο σύστημα. Αυτό γίνεται υπό το συντονισμό του ΟΗΕ όπου έχουν καθοριστεί στάνταρ, βέλτιστες πρακτικέ ε, κτλ. Αλλά ο καθένα πρέπει να καθορίζει τη δική του πολιτική. Και αυτή είναι η δική μα πολιτική εδώ ότι έχουμε πλήρως ανεξάρτητη ε, δυνατότητες από την αγιοστατική τροχιά, κάτι ζωτικό για την προστασία της ζωής και της ιδιοκτησίας και κανείς δεν το κάνει στη θέση σας αυτό, αλλά για την ε, πολική τροχιά δεν μπορούμε να είμαστε πλήρως αυτόνομοι δεν ε, γίνεται οικονομικά αλλά έχουμε κάποια αυτονομία έχουμε έλεγχο του κομματιού του συστήματος που παρέχει μέρος των παρατηρήσεων αλλά ουσιοδών παρατηρήσεων ε, υψηλής αξιοπιστίας και μετά έχουμε και την ε, αντοχή μέσω της Διεθνού συνεργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι για την παγκόσμια γεωσκόψη ούτε οι δεν μπορούν ε, να τα έχουν όλα. Λαμβάνουν περισσότερες προφορές από ό,τι δίνουν. Ας περάσουμε τώρα στην ουσία της σημερινής συζήτησης οι δορυφόροι της UMETSAT είναι διπλής χρήση, όπως γνωρίζετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και του ΝΑΤΟ. Έχουμε την έννοια της ηγέτητος χώρας, έχουμε τυποποιημένα εργαλεία προβλέψεων, ε, ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ στρατιωτικών δυνάμεων. Αν δείτε τον καιρό σε πραγματικό χρόνο, είναι πολύ σημαντικός για την διαχείριση περιφερειακών κρίσεων. Πρέπει να σας πω ότι με ξύπνησαν μέσα στη μέση της νύχτας μια φορά οι Αμερικανοί πριν την ε, εισβολή στο Ιράκ διότι είχε υπάρξει κάποια αμοθίελα και υπήρχε πρόβλημα με κάποιο δορυφόρο και νόμιζαν ότι έφταιγε ο κύριος Βελιπάν επειδή εγώ ήμουν Γάλλος με ρώτησαν ε, έφταιγε ο κύριος Βελιπάν που μίλησε στα Ηνωμένα Έθνη αλλά χρειάστηκε να αναβάλουν για μία μέρα την επίθεση. Ε, είναι απαραίτητο όλες αυτές τι πληροφορίες για την υποστήριξη όλων των επιχειρήσεων. Ε, και έχουμε και ένα πολύ καλό δροφόρο πάνω από τον Ειδικό Ωκεανό, πολύ σημαντικό. Είναι, ε, και τώρα είναι πάνω από τη Συρία. Ε, η πολική τροχιά είναι επίση σημαντική γιατί όπως σας είπα προσφέρει καλές προβλέψεις για ολόκληρο τον κόσμο σε οποιοδήποτε χώρο στρατηγικού ενδιαφέροντος. Λόγω της διπλής χρήση στη UMEDSAT ε, έχουμε τη δυνατότητα να ε, απαγορεύσουμε την πρόσβαση σε κάποια κρίσιμα δεδομένα. Εκπέμπουμε δηλαδή μέσω τηλεοπτικής τεχνολογίας ε, για να διαθέσουμε τα κρίσιμα δεδομένα στην Ευρώπη και αλλού. Αλλά ελέγχουμε ακριβώς οτιδήποτε δίνουμε σε οποιοδήποτε χρήστη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό και είναι και κρυπτογραφημένα τα δεδομένα αυτά. Τώρα, ποιες είναι οι απειλές, ε, οι κυριότερες αντιληπτές απειλές ε, για να φορέα σαν εμάς. Πρώτα απ' όλα τα διαστημικά απόβλητα. Έχουμε έναν ελιγμό κατά μέσο όρο το χρόνο για κάθε ε, ε, ε, δορυφοροπολικής τροχιάς αλλά όλα ξεκινούμε με την υπεύθυνη πολιτική. Συμμορφωνόμαστε με το πρότυπα ISO 24113 και τα κράτη-μέλη μας έχουν συμφωνήσει επίσης για την προηγούμενη γενιά δορυφόρων και υπάρχουν και προειδοποιήσεις που λαμβάνουμε από τις ΕΠΑ, από την JSPOC, διότι έχουμε το ολοκληρωμένο σύστημα, έχουμε υποστήριξη από την JSPOC και τώρα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες SST της Ευρώπης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Ο... Προβλέψεις ε, διαστημικές ε, και ε, μετρολογικές είναι κάτι που χρησιμοποιούμε πολύ αλλά σήμερα οι δορυφόροι είναι πιο ευαίσθητοι στην κοσμική ακτινοβολία και στην ηλιακή δραστηριότητα. Και αυτό που είναι σημαντικό για μας ε, είναι η αντοχή των δορυφόρων μας. Διότι δεν υπάρχει μια υπηρεσία σε πραγματικό χρόνο, αν αυτή η υπηρεσία διακοπεί, ε, πρέπει να διακοπεί για το λιγότερο δυνατό χρόνο. Μια άλλη σημαντική απειλή, όλο και μεγαλύτερη, είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η ασφάλεια των πληροφοριών. Ε, γι' αυτό έχουμε το σύστημα ε, διαχείρισης ε, ασφάλειας πληροφοριών όπως το ISO 27000 δεν είναι απλά ένας κατάλογος ελέγχου, είναι κάτι που εξελίσσεται διαρκώς. Μια άλλη απειλή, λιγότερο προφανής, είναι η πρόσβαση στο φάσμα συχνοτήτων και στις στηρίδες τροχιών. Ο δικός χάρτης 5G, για παράδειγμα, είναι θέμα για μας, γιατί ορισμένε από τις στοχευμένες συχνότητες είναι ε, ε παρατήρηση στο μικροκλιματικό φάσμα για μας ε, και μπορεί να επηρεάσουν και την πρόσβαση στα δεδομένα. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αλλά υπάρχει συντονισμός με την ΕΣΑ, με την Επιτροπή κτλ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και εσείς ε, ως Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλάβετε ότι δεν είναι ότι οι δορυφόροι μας ακόμα και αν δεν είναι στο Κοπέρνικους είναι εξίσου σημαντικοί για τους πολίτες, είναι σημαντικοί για την ασφάλεια των ανθρώπων και ε, των ιδιοκτησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όσον αφορά το περιβάλλον πολιτικής και τις τάσεις Φυσικά πολλά πράγματα γνωρίζουμε. Έχουμε τη φυσική εξέλιξη των συγκρούσεων ότι υπάρχει στο διάστημα. Υπάρχει στο διάστημα και υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για πολλαπλές συγκρούσεις. Επίσης έχουμε κάτι που ζήσαμε ε, ε, πρόσφατα, απομάκρυνση ε, παλαιών δορυφόρων μετρολογικών. Ναι, με απόβλητα ε, σε τροχιά πολύ κοντά στους δικούς μας δορυφόρους, αλλά έχουμε και νέες εξελίξεις, νέες προκλήσεις στην ε, ανάπτυξη πιθανών ε, αστερισμών ελιό, κάτι πιθανό. Και επίσης ε, πολλαπλησιασμό των CubeSat που έχουν μικρή διάρκεια ζωής. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται οι απειλές διαρκώς. Οπότε είναι σημαντικό να υπάρχουν οι σωστές υπηρεσίες προστασίας η του στον κυβερνοχώρο δεν χρειάζεται να επεκταθώ σε αυτήν, θα τη γνωρίζετε καλά. Ε, πρέπει να την παρακολουθούμε προσεκτικά, οι απειλές όλα να εξελίσσονται, όχι μόνο για τους δορφόρους, αλλά και πάνω στη γη. Τώρα δείτε τι γίνεται με την πολιτική, με τα θέματα πολιτικής. Η αμερικανική πολιτική αλλάζει. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα αλλάξει. Ε, ακόμα έχουμε την πολιτική του 2010 του και ο πρόεδρο Ομπάμα λένε σαφέ ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Εμείς έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει μια τάση να ζητείτε περισσότερη αυτονομία παρά ε, αντοχή για, ε, μέσω της συνεργασίας που ήταν το δόγμα της προηγούμενης κυβέρνησης. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα ακόμη. Όταν μιλάμε για τα συστήματα ε, γεωσκόπησης, ε, αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση ε, για το τι θα γίνει, τι υποστήριξη θα δίνεται στους εμπορικούς φορείς. Θα υπάρχει μάλλον μια, ένα σύστημα διτό ένα για δυτικούς φορείς και ένα για τα κράτη. Όλα αυτά αντιστοιχούν σε δισεκατομμύρια επενδύσεων. Επίση, μια νέα τάση είναι η εμπορευματοποίηση του διαστήματος συμπεριλαμβανωμένη τη σελήνη. Και αυτή η εμπορευματοποίηση θα πρέπει να γίνει ε, τηρώντας τις ε, απαιτήσεις ασφαλείας ε, ε των ΗΠΑ. Και εδώ προστίθεται μια νέα διάσταση ε, η αντιπαράθεση μεταξύ της ειρηνικής και της στρατιωτικής χρήσης του διαστήματος. Ε, οπότε ε, θα δημιουργεί το γραφείο της εμπορευματοποίησης του διαστήματος, η διαχείριση της διαστήματης ε, κυκλοφορίας και η εξέλιξη του SSA, κάτι που πρέπει να συζητήσουμε στην Ευρώπη. Τώρα ποια είναι τα ζητήματα για την Ευρώπη. Ας περάσουμε ξανά στο μετρολογικό μοντέλο. Αν δεν υπάρχει άριστο σύστημα, είναι ελάχιστε οι ευκαιρίε αυτονομίας και του να παίξει κανείς σημαντικό ρόλο ε, ώστε να έχει ε, ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ και θέση για ε, τη λήψη δεδομένων που χρειάζεται. Οπότε χρειάζεται η Ευρώπη ένα καλύτερο σύστημα παρατήρησης και ειχνηλάτησης ως θεμέλιο για να μπορεί να συζητήσει με τη ΣΥΠΑ. Για το μετρολογικές εσείς υπάρχει δυνατότητα για ένα μεικτό σύστημα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή αποστολή στο Lagrange 5 και θα μπορούσαμε να έχουμε και διαλειτουργικότητα με τα συστήματα SSA, τον είπα. Είναι σαφέ ότι όπω και στη μετρολογία χρειάζεται κοινή χρήση των δεδομένων για να υπάρχει καλύτερη δυνατή υπηρεσία. Η διαλειτουργικότητα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και τώρα τι γίνεται στο διεθνές πλαίσιο όπου θα είναι όλες οι πληροφορίες χρήσιμες από παντού ε, και τα Ηνωμένα Έθνη είναι κάτι σημαντικό και το SSA τώρα τι θα σημαίνει η εμπορευματοποίηση, ποιες υπηρεσίες θα δίδονται κτλ. Ε, κύριε Πρόεδρε, εδώ ολοκληρώνει την παρουσίασή μου. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρατιέ. Τώρα ο κύριος Φιλίπ Προκρινέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Γενική Διάθεση GROW. Εγώ θα μιλήσω γαλλικά, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε και που είναι και σε μια επίκαιρη στιγμή, γιατί πρόσφατα πέρυσι οθετήσαμε την διαστημική μας στρατηγική και έχουμε διάφορα προγράμματα που ε, υπόκειται σε αξιολόγηση. Οπότε πολύ σύντομα θα ξανάρθουμε στο Συμβούλιο και την Επιτροπή για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του επόμενου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Και φυσικά θα χρειαστεί η υποστήριξή σας. Χαίρομαι για την πρόσφατη έκθεση για την ε, διαστημική στρατηγική. Αρμόδια κατ' ουσία είναι η Επιτροπή Ήτρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για την συνεισφορά σας ε, που σχολιάζει διάφορα τμήματα αυτής της στρατηγικής. Στα πλαίσια της ε, διαστημικής μας στρατηγικής οι πιο σημαντικοί στόχοι που ενδιαφέρουν και τη σημερινή συζήτηση είναι να εξασφαλίσουμε στην Ευρώπη αυτόνομη πρόσβαση και ασφαλή πρόσβαση στο διάστημα. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι εκ των για να εξασφαλίσουμε καταρχήν την αυτονομία της Ευρώπης και την αυτόνομη πρόσβαση σε κάποια τεχνολογικά μέσα, αφενός και αφετέρου, ε, επιτρέψουμε στους Ευρωπαίους πολίτες να επωφεληθούν από τις συνέπειες των δραστηριοτήτων μας στο διάστημα. Ο Αλέα Ρατιέ μας έδωσε ένα παράδειγμα διαστημικής υποδομής που συνδυάζει και στρατιωτικά και μη στρατιωτικά πολιτικά συμφέροντα. Μάλιστα τα περισσότερα προγράμματα, είτε το Γαλλιλαίο είτε το Κοπέρνικος, το Γαλλιλαίο είναι πιο άμεσο γιατί με το, την υπηρεσία PRS έχουμε μια υπηρεσία που έχει μια πτυχή ασφάλειας και μάλιστα και στρατιωτικής και με το Κοπέρνικος έχουμε την υπηρεσία της ασφάλειας και μία από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να ε, εκμεταλλευτούμε, να εξορθολογήσουμε και να καταστήσουμε πιο αποτελεσματική τη χρήση του Κοπέρνικους για να ενισχύσουμε την πτυχή της ασφάλειας πολιτικής ή στρατιωτικής. Και όταν μιλώ για πολιτική ασφάλεια ή πολιτική προστασία, εννοώ κυρίως ε, την ε, επιτήρηση των συνόρων. Επίσης, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια σφαιρική προσέγγιση και έποψη ε, αυτής της διτής χρήσης, που είναι ταυτόχρονα στρατιωτική και μη στρατιωτική πολιτική. Και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης της Άμυνας που πρόσφατα υιοθετήσαμε και των συζητήσεων που θα γίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πρώτο βιομηχανικό πρόγραμμα με ανάπτυξη ικανοτήτων που θα συνδυαστεί με ένα ερευνητικό πρόγραμμα θα δούμε τα όρια μεταξύ των ερευνητικών προγραμμάτων διαστημικής έρευνας ε, που θα αφορούν την άμυνα και που σε κάποιους τομείς θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Γιατί μιλήσαμε για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έχει σαφώς μία στρατιωτική ε, ε, διάσταση, αλλά και μία διάσταση πολιτικής προστασίας ή ασφάλειας πολιτικής. Και τα δύο προγράμματα, και το Κοπέρνικος και το Γαλιλαίο, πάνε μια χαρά. Η πρώτη υπηρεσία του Γαλιλαίου ξεκίνησε πέρσι το Δεκέμβριο και προβλέπεται να ανακτήσει την πλήρη επιχειρησιακή του ικανότητα το 2020 το πρόγραμμα Γαλιλαίος. Σε ό,τι αφορά τις ε, ε, του Κοπέρνικους, τα Sentinel, συνεχίζεται η ανάπτυξη όπως, είχε, όπως προβλεπόταν και το θέμα της ασφάλειας έχει ανατεθεί σε τρεις διαφορετικούς φορείς. Το Κέντρο Δορυφόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΣΑΤΣΕΝ, μάλιστα είχατε ακρόαση με τον Γενικό Διευθυντή του πρόσφατα, τον κύριο Λεγκέ. Τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής, το Frontex, για την ε, ασφάλεια στη θάλασσα, την ΕΜΣΑ που εδρεύει στην Λισαβόνα. Αυτή είναι οι τρεις φορείς. Και μάλιστα δεδομένου ότι ο Κοπέρνικος, παρόλο που δεν το γνωρίζουν πολύ, ήταν και εξακολουθεί να είναι ε, ο βασικός μας πελάτης anchor customer, όπως τα λέμε στα αγγλικά, ή ο πρωταρχικός χρήστης ε, του συστήματος DRS που επιτρέπει στους δορυφόρους τη μεταξύ τους επικοινωνία, ώστε να μην ε, περιμένουμε να ξαναβρούμε από τις κεραίες μας τον δορυφόρο για να έχουμε πρόσβαση στο σύστημα. Αλλά χάρη στην ανταπόκριση μεταξύ των δορυφόρων μπορούμε να έχουμε ανα πάση στιγμή πρόσβαση στα δεδομένα. Και μάλιστα επειδή είναι κρυπτογραφημένο το σύστημα, είναι ένα ιδανικό σύστημα για την μεταβίβαση δεδομένων, ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών. Επίσης, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στο Κοπέρνικους και για την ασφάλεια θα αναπτύξουμε και τις μη διαστημικές παρατηρήσεις, όπως λέγονται. Γιατί όλο και πιο συχνά ε, ο οργανισμός Frontex αναφέρεται στην ταυτόχρονη χρήση των δεδομένων που λαμβάνουν οι δορυφόροι και των δεδομένων που λαμβάνουν τα drones, τα μη επαδρομένα μικρά σκάφη. Και μάλιστα ε, ε, προτάθηκε και η δημιουργία πλατφορμών ε, άνω της ε, στρατόσφαιρας, οπότε σκόπιμο είναι να έχουμε ένα ανοιχτό σύστημα, γιατί για την παρατήρηση της γης, ε, για τη γεωσκόπηση δεν έχουμε ποτέ ένα τέλειο σύστημα. Όσο περισσότερους πομπούς έχουμε, τόσο, ελίπτες έχουμε, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το σύστημα. Ε, φυσικά περιοριζόμαστε και από τους νόμους της φυσικής. Οπότε εξορισμού ένα τμήμα είναι η αγορά δεδομένων για τον απλούστατο λόγο ότι λαμβάνουν χώρα κάποια γεγονότα που δεν είναι εύκολο να τα παρακολουθούμε συνέχεια με τη χρήση των δορυφόρων. Τώρα, για τα θέματα της ασφάλειας, κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει η συζήτηση ώστε για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να προτείνουμε την πρωτοβουλία GovSatCom, δηλαδή ε, δορυφόρους για τη δορυφορική επικοινωνία με δεδομένα που θα διαχειρίζονται θεσμικά όργανα. Οπότε θέλουμε αξιόπιστους και θεκτικούς δορυφόρους που θα περι... επιτρέπουν εκτεταμένη χρήση. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, σε αυτές ε, τις επικοινωνίες ε, για κυβερνητική χρήση, έχουμε, θα έχουμε όλο και περισσότερες ανάγκες για τις κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες και κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα κρίσιμο κατόφλι. Για παράδειγμα, και εδώ άσχετα αν μιλούμε για στρατιωτική ή μη στρατιωτική χρήση ή μόνο για, για πλήρη πολιτική χρήση. Όλοι μιλούμε για την ανάπτυξη των drones υψηλής ε, σε μεγάλο ύψος και μάλιστα ε, τα, οι δορυφόροι συμπληρώνουν τα drones και το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο γιατί οι δύο πυλώνες που μας επιτρέπουν την ασφαλέστατη και αξιόπιστη χρήση των drones, των μη επανδρομένων σκαφών, είναι να έχουμε καταρχήν επικοινωνία ευρυζωνική, γιατί θα πρέπει τα ντρόνα να μπορούν να μα μεταβιβάζουν τι πληροφορίε που συγκεντρώνουν και επίσης ε, να δίνονται εντολέ που θα πρέπει να είναι υπεράνω των ε, δράσεων κάποιων κακόβουλων φορέων. Οπότε η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι δεύτερο πυλώνα τη αποτελεσματικότητα των drones. Και σε ό,τι αφορά το GovSatcom, τι κυβερνητικέ δορυφορικέ επικοινωνίε, πέραν των drones, έχουμε και πολλέ άλλε χρήσει. Στρατιωτικέ ή μη. Και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάναμε ε, έναν εξονυχιστικό έλεγχο και επισκόπηση όλων των αναγκών, των πολιτικών αναγκών και ζητήσαμε α, αντίστοιχη μελέτη και από τον οργανισμό και καταλήξαμε σε μία ανάλυση επιπτώσεων αντικτύπου που θα είναι έτοιμη στα τέλη του χρόνου. Οπότε θα ακολουθήσει κατά πάσα πιθανότητα μετά από αυτό μια νομοθετική πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια, πλαίσια των νέων προγραμμάτων και νομικών βάσεων για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπω θα διαπιστώσατε, στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο δεν υπάρχει μια δημοσιονομική γραμμή για τέτοια πρωτοβουλία, παρά μόνο στο πρόγραμμα ερευνών Ορίζοντα 2020. Και φυσικά υπάρχει και το πρόγραμμα SST. Θα σας ε, μιλήσει και ο κύριος Ντένσινγκ αργότερα. Το ανέφερε και ο κύριος ε, Ρατιέ. Πρόκειται για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την επιτήρηση και παρακολούθηση των αποβλήτων του διαστήματος. Και έχει ξεκινήσει από τα μέσα του 2015 και οι αρχικές του υπηρεσίες ήδη παρέχονται από την 1η Ιουλίου 2016. Μία θεσμική παρατήρηση τώρα θα παρατηρήσατε ότι αυτό το πλαίσιο του συντονισμού δεν είχε προβλεφθεί στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο του, που ψηφίστηκε το 2013. Οπότε έπρεπε να τροφοδοτήσουμε το πρόγραμμα SST με μία μεταφορά κονδυλίων κυρίως από το πρόγραμμα Γαλιλαίο ή από τον ορίζοντα 2020 και το Κοπέρνικο. Τι γίνεται με το πρόγραμμα λοιπόν αυτό της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος. Ε, ήταν κάπως ε, προβληματική η έναρξή του, γιατί στο ισχύον πλαίσιο απαιτείται διακυβερνητική συνεργασία βάσει κριτηρίων μεταξύ των χωρών που έχουν τη σχετική ικανότητα. Γιατί ξέρετε ότι η διακυβερνητική συνεργασία δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα στις Βρυξέλλες. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα που φυσικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να δούμε τι είδου βελτιώσει επιδέχεται το σύστημα και να τι προτείνουμε για το επόμενο πολίτε δημοσιονομικό πλαίσιο. Καταρχήν, γιατί θέλουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Γιατί εξαρτώμαστε απόλυτα μέχρι στιγμή από το αμερικανικό. Και δεν είμαστε σίγουροι ότι το αμερικανικό σύστημα θα συνεχίσει ε, δωρεάν να μας παρέχει στοιχεία και δεδομένα ή θα συνεχίζει να μας τροφοδοτεί όπως έκανε μέχρι τώρα. Απ' την άλλη πλευρά, ένα τρίτο των παγκόσμιων δορυφόρων είναι ευρωπαϊκοί. Και μεταξύ τους έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το, θα έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2020, αν προσθέσουμε και το Κοπέρνικος και θα έχουμε περίπου 40 δορυφόρους σε τροχιά. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ένωση ε, κρατών μελών που καλύπτει τα, τις ανάγκες και των ε, ευρωπαϊκών φορέων, ένα τρίτο των παγκόσμιων δορυφόρων, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 40. Οπότε έχουν, υπάρχει η ανάγκη για αυτόνομο δικό μας σύστημα, ανεξάρτητο. Και σιγά σιγά θα πρέπει στα πλαίσια του συστήματος να βελτιώσουμε την ισχύουσα διακυβέρνηση μετά την εμπειρία που θα αποκομίσουμε και επίσης να επικαιροποιήσουμε και να αναβαθμίσουμε το σύστημα ώστε να αποκτήσουμε σταδιακά αυτή την αυτονομία απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ε, δεν θα μας χρειάζονται πια τα αμερικανικά δεδομένα. Γιατί μακροπρόθεσμα ε, μια και τα συστήματα θα γίνονται πιο απαιτητικά από τεχνολογική άποψη και πιο δαπανηρά και πιο πλήρη γιατί αρχικά μιλούσαμε για την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος, το SST, αλλά θέλουμε να βελτιώσουμε και να διευρύνουμε και την πρόβλεψη του διαστημικού περιβάλλοντος, όπως μας είπε πριν ο Άλλα Ρατιέ, ε, στα πλαίσια του SSA. Και επίσης, ε, να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι να προβλέψουμε τον κίνδυνο σύγκρουσης ε, ε, δορυφόρου μεταξύ τους ή σύγκρουσης κάποιων φυσικών ε, αντικειμένων με τη γη. Οπότε θέλουμε να διευρύνουμε το SST για να καλύψουμε και την, τον καιρό του διαστήματος, το διαστημικό περιβάλλον, να, έχουμε μια, να βελτιώσουμε το SSA, την ενημέρωση της κατάστασης του διαστήματος, για να αποφύγουμε την ε, σύγκρουση της γης με αντικείμενα επίσης και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια κατάλληλη λειτουργία, εύρυθμη λειτουργία του SST, της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος και θέλουμε εδώ δύο βασικές βελτιώσεις. Καταρχήν βελτίωση των ικανοτήτων που ήδη έχουν κάποια κράτη-μέλη, όχι όμως ε, ε, να καταλήξουμε στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή μόνο μεταξύ των διαφόρων συστημάτων. Το σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος δεν είναι μέσο εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων. Γιατί ακριβώς επειδή τα εθνικά συστήματα ήταν αποτελεσματικά έχουν πρόσβαση στο SST. Οπότε τα πέντε κράτη που συμμετέχουν στο SST θα πρέπει ε, να κάνουμε μια ευθυγράμμιση προς τα πάνω και όχι μια ευθυγράμμιση προς τα κάτω. Και κάτι άλλο που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι η θέση των δεδομένων σε δίκτυο. Η Ευρωπαϊκή όμως Επιτροπή ε, δεν μπορεί να είναι βέβαιη για την εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών των κρατών μελών. Γιατί αν στο στη σύμπραξη αυτή δεν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποφεληθεί από τις, ε, την τροφοδοσία με δεδομένα από δύο χώρες που μεταξύ τους δεν έχουν σχέσει ή δεν έχουν εμπιστοσύνη. Οπότε στα πλαίσια του SST θα πρέπει να ελέγξουμε πρώτα τις τεχνικές πτυχέ και τις πτυχέ ε, τροφοδότηση του συστήματος του δικτύου. Επίση ε, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη διακυβέρνηση, γιατί αυτό είναι ένα αίτημα και των κρατών μελών και θα χρειαστούν και κάποιες αλλαγές στην οτροπία κάποιων κρατών μελών ώστε να αντιληφθούν τα κράτη-μέλη ότι όπως είπε και ο κύριος Ρατιέ, το SST όπως και άλλα πολλά ευρωπαϊκά συστήματα διαστημικά ε, έχουν ευρωπαϊκό επίπεδο για τον απλούστατο λόγο ότι το απαιτούμενο επίπεδο δεν μπορεί να υλοποιηθεί από κανένα κράτος μέλος μεμονωμένα. Χωρίς συντονισμό λοιπόν δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Και τέλος, και εδώ θα ολοκληρώσω, το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, που είναι πανταχού παρούσα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα πλαίσιο για τις υβριδικές απειλές, τώρα το δρομολογούμε, και οι υπηρεσίες της ε, Γενικής Διεύθυνσης GROW ασκούν ένα συντονιστικό ρόλο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε 10-12 γενικές διευθύνσεις που συμμετέχουν σε αυτό το σχέδιο δράσης. Θα εκπονήσουμε μάλιστα και έκθεση στις 19 Ιουλίου, την επόμενη εβδομάδα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε για το διάστημα αν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ε, πρέπει να ληφθούν και συμπληρωματικά μέτρα για το διάστημα. Κάθε φορά που έχω την ευκαιρία και την τιμή να έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα επαναλάβω κάτι που λέω συνήθω και που είναι λογικό για κάθε υπάλληλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα προετοιμάσουμε ήδη και τη συνέχεια των εφισταμένων προγραμμάτων για το επόμενο ΠΔΠ. Φυσικά το διάστημα είναι μια δαπανηρή διαδικασία, ένα δαπανηρό εγχείρημα και έχουμε ένα είδο δαπανών που είναι σχεδόν υποχρεωτικέ. Δηλαδή δεν μπορούμε να σταματήσουμε κάτι που έχουμε ήδη ξεκινήσει. Θα είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τα μέχρι τώρα προγράμματα. Οπότε ε, για τα διαστημικά προγράμματα αλλά και για τα προγράμματα άμυνα θα υπάρχει ένα πυρήνα αναγκών που δεν θα επιδέχεται περικοπέ. Οπότε το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι αυτό που θα περιλαμβάνει τις σχεδόν υποχρεωτικές δαπάνες λόγω των ήδη ε, ε, ε, εφαρμοσμένων προγραμμάτων. Και αυτό δεν μπορούμε να το συμπιέσουμε με τίποτα, αυτό το, αυτές τις δαπάνες, αυτό τον πυρήνα. Οπότε για να αξιοποιήσουμε τις προηγούμενες επενδύσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνέχειά τους και αυτή η συνέχεια θα είναι δαπανηρή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Από την ΕΖΑ τώρα, ο Διευθυντής κύριος Ντάντζιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που με προσκαλέσατε να δώσω μαρτυρία ενώπιον της Επιτροπής σας σήμερα. Επιτρέψτε μου να σας ε, θυμίσω ότι πριν από ένα περίπου χρόνο ήταν εδώ παρόν ο Γενικός μας Διευθυντής για να σας ενημερώσει για τις δραστηριότητες ασφαλείας της ΕΖΑ σε γενικού όρου. και μια και έχω εγώ την αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Κέντρου ε, της ΕΖΑ θα ε, ήθελα σήμερα να σας μιλήσω συγκεκριμένα για την προστασία των διαστημικών υποδομών που είναι το θέμα της ε, σημερινής σας διάσκεψης. Η έκθεση στην οποία υπόκεινται οι υποδομές του διαστήματος σε επιθέσεις διαφόρων είναι πραγματική. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός. Και ας κοιτάξουμε κάποια δεδομένα. 750.000 κομμάτια συντριμιών διαστημικών με μέγεθος ε, ανώτερο του ενός ε, εκατοστού είναι σε κίνηση. Και αυτό σημαίνει από ένα εκατοστό μέχρι μεγέθου δορυφόρου, γιατί έχουμε χιλιάδες δορυφόρους σε κίνηση στο διάστημα αυτή τη στιγμή. Από ένα σημείο και μετά ε, ε καθίστανται ανεξέλεγκτοι και άρα συνιστούν πολύ σημαντικό και συγκεκριμένο κίνδυνο. Επίσης, θα υπενθυμίσω πως βρισκόμαστε στην, ε, ε, στις αρχές της εκτόξευσης υπερ διαστημικών συστημάτων, ε, υπερμεγεθών, υπερμεγεθών μάλλον διαστημικών συστημάτων. Έχουμε από μια κυβέρνηση, παραδείγματι από μια χώρα, την ανακοίνωση ταυτόχρονης εκτόξευσης 600 δορυφόρων και αυτό θα το ακολουθήσουν και άλλες και άρα ε, έχουμε σημαντική ενίσχυση των διαστημικών συντριμιών και αποβλήτων στο διάστημα και βέβαια πρέπει να διαφυλαχθεί η ε, βιωσιμότητα του διαστήματος και για τις επόμενες γενναίες. Αυτό είναι το δικό μας καθήκον. Επίσης, ε, η διαχείριση της κυκλοφορίας του διάστημα, όπως ακριβώς και η διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας. Έχουμε να κάνουμε με μια καθημερινή δραστηριότητα βέβαια στα αεροδρόμια και σα είναι γνωστή, αλλά αντίστοιχα και η διαστημική κυκλοφορία πρέπει κάπω να διαρρυθμιστεί, να ρυθμιστεί. Πολύ πιο ο βέβαια να μπορέσει κανεί να υπολογίσει την πορεία ενό αεροπλάνου που ξεκινάει το πρωί, απογειώνεται, μετά προσγειώνεται από κάποιε ώρε. Δεν υπάρχει τίποτε το διαφορετικό σε κάθε τέτοια πτήση, ενώ στο διάστημα έχουμε πολύ διαφορετικέ συνθήκε και πρέπει κάπω να ρυθμίσουμε το περιβάλλον γύρω από εμά, Το ευρωπαϊκό λοιπόν πολεμικό Κέντρο εδώ και 50 χρόνια και μάλιστα φέτος γιορτάζουμε την 50η μας επέτειο, διαχειρίζεται διαστημικούς δορυφόρους ε, και βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια και τις δεκαετίες συλλέξαμε γνώσεις σε σχέση με το διαστημικό περιβάλλον και γι' αυτό ε, είναι ανεγνωρισμένο το γραφείο διαστημικών συντριμιών ως ε, αρχή παγκοσμίου, παγκοσμίου κύρους ως προς την αντιμετώπιση των κινδύνων από την έσοδο, είσοδο ε, στην ατμόσφαιρα ή τον κίνδυνο εισόδου στην ατμόσφαιρα συντριμιών. Όπως είπαμε λοιπόν, Ω προ τη διαχείριση τη βάση δεδομένων, ω προ τη βάση δεδομένων για τα διαστημικά συντρίμια, εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό από του εταιρούς μα των ΗΠΑ και ναι, θα το ομολογήσω ότι του φθονούμε κατά κάποιο τρόπο, αλλά ταυτόχρονα χαιρόμαστε ιδιαίτερω και είμαστε ευγνώμονε για το γεγονό ότι μοιράζονται μαζί μα αυτέ τι πληροφορίε πληροφορίες ο Γενικό Μεθοδητής, αλλά και εγώ ίδιο υποστηρίζουμε ιδιαίτερω την, ε, το άνοιγμα των γνώσεων, δηλαδή την ε, αμοιβεοποίηση των γνώσεων που συλλέγουμε ως προς τα διαστημικά συντρίμια σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό βέβαια για μας θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί τελικά όλοι μέσα στην ίδια ε, βάρκα βρισκόμαστε, όλοι θέλουμε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε διαστημικά οχήματα με τρόπο ασφαλή χωρίς κίνδυνο σύγκρουσης. Άρα λοιπόν όσοι έχουν μεγαλύτερη διαχείριση διαστημικών οχημάτων θα υποφεληθούν και περισσότερο από αυτήν την ε, αμοιβεοποίηση των γνώσεων όπως είναι άλλωστε και υπεύθυνοι για, ε, για τον πολλαπλασιασμό των διαστημικών συντριμιών. Άρα, αυτή, αυτό το πνεύμα της ε, κοινότητα και συνεργασίας που ήταν γνωστό από το σύστημα Γαλιλαίος, μας το εξέτασε νωρίτερα ο προηγούμενος ομιλητής, ε, το βλέπουμε και εδώ. Και ξέρετε όταν ετοίμαζα την ε, ομιλία μου για να έρθω εδώ, προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να διατυπώσω κομψά τα διάφορα ζητήματα που άλλωστε με πολύ μεγάλη επιτυχία περιέγραψε ο κύριο Μπριουνέ, τα ζητήματα δηλαδή τη διακυβερνητική συνεργασία, την απουσία τη εναρμόνιση ε, των συστημάτων και την έκκληση για άρση όποιων εμποδίων σε ε, εσωτερικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μπορεί να απευθύνουμε εκκλήσει για παγκόσμια συνεργασία, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε κι εμεί ότι στο εσωτερικό μα δεν έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε. Μπορεί να έχουμε κοινού πόρου για πράγματα ε, που κάνουμε, αλλά δεν έχουμε λύσει απλά προβλήματα όπως το, τα διαστημικά συντρίμια και απόβλητα. Ο Γενικό Διευθυντή τη HumanSat μα μίλησε για την διαστημική ύλη και μια πιθανότητα για κοινή πρωτοβουλία που είναι υποπρογραμματισμό αυτή τη στιγμή με τους εταίρου μας από τις ΗΠΑ, τη ΝΟΑ. για τη διαστημική ύλη όπως και για την διαστημική ε, ανείχνευση και ιχνηλασία. Και σε αυτό θα πω ότι ναι, βεβαίω είμαστε ευγνώμονε για τη δυνατότητα συνεργασία, αλλά ω προ τη βάση δεδομένων δεν έχουμε ε, ρυθμιστικό πλαίσιο. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί εταίροι μα προηγούνται. Θα ήταν πολύ καλύτερο να μπορούσαμε κι εμεί να έχουμε κάτι τέτοιο για να ξέρουμε σε ποιο. Ε, σε ποια τροχιά θα κυκλοφορήσουν οι δορυφόροι μας, ώστε να μην μας το επιβάλλουν αυτό οι εταίροι, αλλά να έχουμε εμείς τους δικούς μας κανόνες. Άρχισα λοιπόν τις επαφές με τους Αμερικανούς εταίρους ε, σε μια κοινή αποστολή για την αντιμετώπιση των ε, διαστημικών των ζητημάτων διαστημικής ύλης. και μου είπαν ότι μπορούν να έχουν ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα απόσταση με το, το σύστημα που μετράει σε τέτοιες μονάδες, απόσταση από τη γη προς τον ήλιο ε, τροχιά, αλλά σε πολύ πιο κοντινή τροχιά θα έχουμε τη μετεωρολογική παρατήρηση και αντίστοιχα την αμοιβαία ενημέρωση. Άρα οι αποστολές, οι αμερικανικές αλλά και οι ευρωπαϊκές, θα συνεργάζονται, θα ανταλλάσσουν δεδομένα και χαίρομαι γιατί αυτό είναι μια ιδέα η οποία θα μας οδηγήσει σε ένα πολύ στέρεο σύστημα για την κοινή αξιοποίηση των, ε, του δυναμικού που έχουμε στο διάστημα. Είχαμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση το 2003 και αυτή ήταν η απαρχή με 46 καταγραφές ζητημάτων από 70 που συζητήθηκαν διεξοδικά και μας ε, βοήθησαν στην περαιτέρω συνεργασία. Επίσης, Στις επενδύσεις ε, έχουμε όφελος προφανώς από τη συνεργασία με συντελεστή μόχλευσης 6 εξαπλασιάζουμε δηλαδή την απόδοση των επενδύσεών μας. Επίσης έχουμε ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από το 2005, ξεκίνησε σε πολύ, μικρές, σε πολύ μικρή κλίμακα γιατί ήταν μάλλον διστακτικά τα κράτη-μέλη ως προς την ανάπτυξη επενδύσεων στο πρόγραμμα αυτό. Έχει όμως τώρα διπλασιάσει το νόγκο του στην τελευταία υπουργική διάσκεψη του 2016 εκφράστηκε υποστήριξη προς το πρόγραμμα μας με διπλασιασμό της πρικοδότησης και νομίζω ότι αυτό το καθιστά το σημαντικότερο σε όγκο πρόγραμμα και έχουμε τρεις πτυχές στο πρόγραμμα αυτό, παρατήρηση των αντικειμένων που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια της γης, τη μετεωρολογική πρόβλεψη και τα ή μετεωρολογική ύλη απόβλητα συντρίμια. Ειδικά για την πρώτη περίπτωση των εγκύτερων στην επιφάνεια της γης αντικειμένων είναι πολύ σοβαρός ο λόγος της παρατήρησης και συνιστούν μεγάλο κίνδυνο και πρέπει να είμαστε σε θέση και να προβλέπουμε κατά το βαθμό του δυνατού την πιθανότητα πτώσης, τον εντοπισμό του σημείου πτώσης και του οδούν κίνδυνο. Είχαμε παραδείγμα το 2002 ε, ένα κομμάτι μετεωρίτη που πέρασε στα βόρεια Ουράλια, κοντά στο Τσίλιαμπίνσκ, πέρασε από την ε, ατμόσφαιρα και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι πέρασε ε, κοντά σε μια αεροκατοικημένη μεν πόλη, αλλά με εφταπλάσια από μια μεγάλη πυρηνική βόμβα ισχύ, ευτυχώς περνώντας από την μπαίνοντα στην ατμόσφαιρα διασπάστηκε σε πολλά μικρά κομμάτια και παρά το γεγονό ότι ήταν όπω είπα αεροκατοικημένη η περιοχή κατεγράφησαν πάνω από χίλια ε, χίλιοι τραυματισμοί, μικροτραυματισμοί από τα θράψματα αυτά. Καταλαβαίνετε δηλαδή ε, αν ήταν διαφορετικέ συνθήκε, πόσο διαφορετικά θα ήταν οι συνέπειε και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε όσο δυνατόν πιο, πιο ακριβή παρατήρηση και βέβαια πρόγνωση, προβλέψει και προειδοποίηση αν και προς το παρόν αυτό που κάνουμε νομίζω δεν ξεπερνά την ε, ε, ορνηθολογία παρατήρηση άγριων πτηνών λίγο πολύ. Θέλουμε να βελτιώσουμε δηλαδή πολύ περισσότερο τις επιδόσεις μας. Και θέλουμε για το μέλλον πιο έντονο χαρακτήρα ευρωπαϊκό στη δουλειά μας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Διαστήματος ΕΟΔ έχει πολλά να προσφέρει κάνουμε καλά τη δουλειά μας και πάνω απ' όλα μπορούμε, και αυτή είναι, αυτός είναι ο ρόλος μας, να ε, υπερκεράσουμε μια κατακαιρματισμένη προσέγγιση που μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Uh, gentlemen, thank you very... Αξιότιμοι κύριοι, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος ε, για αυτές ε, τις ε, παρουσιάσεις, τις εισαγωγικέ και δίνω τώρα το λόγο στα μέλη για τη συζήτηση. Ε, νομίζω ότι ο κ. Στρογεύς και ο συζητητής θα πρέπει να είναι ο που θα μιλήσει για το θέμα αυτό. E, Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμάτα τους τρεις καλεσμένους μας και ε, πραγματικά μένουμε πολύ ικανοποιημένοι από την πρόοδο των εργασιών ε, για τα δορυφορικά συστήματα, για το Κοπέρνικο, στο Γαλιλαίο, αλλά και άλλες δράσεις που συνδέονται με άλλα προγράμματα. Έχω μία ερώτηση και μία πρόταση και μία δεύτερη ερώτηση μετά. Ε, αφορούν κάπως διαφορετικά θέματα. Καταρχήν έχω συνεχώς την ε, αίσθηση ότι δεν γίνονται επαρκείς προσπάθειες για την πρόθεση το, του έργου σας. Δεν προβάλλεται αρκετά το έργο σας. Ε, τα προγράμματα αυτά τα ξέρουν μόνο οι δήμονες ή κάποιοι κυβερνητικοί φορείς και θεσμοί. Αλλά για να βρεθούν ε, τα τεράστια κονδύλια που απαιτούνται για τέτοια έρευνα θα πρέπει να ενισχυθούν τα προγράμματα προώθησης, προβολής, ενημέρωσης και για τις ε, υπηρεσίες που προσφέρουν αυτά τα προγράμματα, για την πρόσβαση. Θα πρέπει αυτά τα ενημερωτικά προγράμματα να έχουν ευρύτερη κάλυψη για να φτάσουν σε περισσότερο κόσμο. Δεύτερο θέμα. Ε, ετησίως, ε, πόσοι δορυφόροι μέχρι τώρα λειτουργικοί πεθαίνουν κατά κάποιο τρόπο, αποσυνδέονται και δεν προσφέρουν πια τις λειτουργίες τους. Ποιος είναι ε, ο βαθμός θνησιμότητας, αν θέλετε, των δορυφόρων και πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτή την ε, ε, διακοπή λειτουργία των δορυφόρων για να μειώσουμε το κόστος. Φυσικά θα πρέπει να ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσουμε την απειλή για τους ενεργούς δορυφόρους των ανενεργών. Ευχαριστώ. Κύριος Γκάλερ. Äh, Ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες ε, ομιλίες σας, για την ενημέρωση. Με εντυπωσιάζουν όλα αυτά που έχουμε καταφέρει όλα αυτά που γίνονται σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα στην άμυνα και την ασφάλεια. Διερωτώμαστε βεβαίως τι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερο από αυτή την ε, συνεργασία. Μιλήσατε για ασφαλή πρόσβαση στο διαστημικό χώρο. Κάτι το οποίο κάνουμε και στον χώρο της πολιτικής προστασίας βεβαίως, αλλά και στο στρατιωτικό τομέα θα μπορούσαμε να κάνουμε αρκετά. Και νομίζω ότι και, στο, και το Γαλιλαίος μας έχει επισημάνει ότι έχουμε σύστημα καλύτερο από ότι οι Αμερικανοί φίλοι μας. Το PRS συγκεκριμένα, που δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνουν ως αρχικά, Επίσης είπατε ότι αναπτύσσεται ένα σύστημα GovSat ε, ε, διακυβερνητικών, κυβερνητικών ε, δορυφορικών τηλεπικοινωνιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά κρατικές αρχές. Μήπως είναι λίγο νωρίς σε σχέση με το Γαλιλαίο και το κόστος ενός τέτοιου συστήματος που έχουμε συζητήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ε, να καλυφθεί μόνο από τον πολιτικό τομέα, τον τομέα της πολιτικής προστασίας, γιατί οι Αμερικανοί το έχουν κάνει διαφορετικά. Έχουν κοιτάξει και την πολιτική διάσταση των στρατιωτικών τους επενδύσεων, ενώ εμείς κάνουμε το αντίστροφο. Ξεκινούμε με την πολιτική προστασία για να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα επέκταση στο στρατιωτικό τομέα. Νομίζω ότι θα έπρεπε αυτό να το κοιτάξουν πιο προσεκτικά αν υπάρχει δυνατότητα για στρατιωτικές χρήσεις και σε αυτό σας ρωτώ εάν ε, υπάρχει κάποια εξέλιξη, πόσες ή ποιες κυβερνήσεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Για την ΕΖΑ. 50 χρόνια εμπειρίας από την ε, λειτουργία δορυφόρων. και την ε, πρόταση για ένταξή τους σε ευρωπαϊκές υποδομές. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι είναι διαφορετικά τα κρατημέλη, διαφορετικές η οργανώ... Ε, διαφορετική οργάνωση, η χρηματοδότηση σε κάθε περίπτωση. Αλλά όπου υπάρχουν δορυφόροι, δομές, επενδύσεις, γιατί να κάνουμε δύο και τρεις φορές το ίδιο πράγμα γιατί νομίζω θα έπρεπε να εκφραστεί πολιτικά η βούληση, μια μια συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και ΕΖΑ, ώστε δυνατόν ε, βέλτιστη δηλαδή αξιοποίηση των υφισταμένων υποδομών της τεχνογνωσία. Και νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό. Ίσως λοιπόν θα ήταν καλό οι δύο από τους ομιλητές μας ε, που αφορά αυτή η πρόταση να μας απαντήσουν. Ο κύριος ε, Γκέμεκαν δεν και δεν είμαι σίγουρη ότι ζήτησε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά τους καλεσμένους μας για τις πληροφορίες που μας έδωσαν, που είναι φυσικά ενδιαφέρουσες. Και θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το αναμενόμενο Brexit, την έξοδο της ε, Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα διαμορφωθούν ε, οι σχέσεις με, τις, ε, με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι και το πιο σημαντικό θέμα η, διαστημική στρατηγική στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του Brexit, αλλά καλό θα ήταν να το έχουμε και αυτό υπόψη. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τις ε, τεχνικές προοπτικές του συστήματος. Το, το σύνολο του συστήματος στηρίζεται σε εννέα δορυφόρους που έχουν ε, την τεχνική τους ε, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Ποια είναι τα σχέδια για την αντικατάσταση ενός τμήματος τουλάχιστον αυτών των δορυφόρων, των νέων δορυφόρων στο μέλλον. Και επίσης, ε, ποιο είναι το κόστος μιας τέτοιας αντικατάστασης. Ευχαριστώ κύριος Βανόρντεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους, πολύ ενδιαφέρουσες. Για το Brexit, ε, αυτή είναι και η αξία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, πιστεύω. Ότι εκεί έχουμε μια δομή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει τη δυνατότητα στο Ενωμένο Βασίλειο να συνεχίσει να συμμετέχει ε, σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ε, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα σαν αυτά. Θα ήθελα όμως να ακούσω και το δικό σας σχόλιο γι' αυτό. Ε, κάτι σχετικό κατά κάποιο τρόπο θα με ενδιαφέρει η δημοσιονομική πτυχή ε, που συζητήσατε. Ποιε θα είναι οι δημοσιονομικές σα ανάγκε ε, για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, σε σχέση με το crowdfunding. Έχετε κάποια ιδέα και πώς θα σχετίζεται αυτό με τη συμβολή σας, με την οικονομική σας συμμετοχή ε, Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ε, ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Έχω και άλλη μια ερώτηση για το ζήτημα της ασφάλειας. Ε, ε, ανησυχείτε καθόλου για τις εξαγωγές ευαίσθητης διαστημικής τεχνολογίας και για τις συνέπειες για την ασφάλεια οποιονδήποτε συμφωνιών εταιρική σχέση που έχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο που να έχει ζητήσει το λόγο, οπότε θέλω να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Oh yeah. I'm, I'm sorry. Ζητά συγγνώμη, Πρόεδρος, το μέλος της Ήτρε, ε, κύριο Κάπελ. Κάπελ, ναι, Πρόεδρε, και εμείς η Επιτροπή Ήτρε ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερως ε, για, το, η για τις εξελίξεις ε, στα διαστημικά θέματα και γι' αυτό και ήρθα άλλωστε, γιατί πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το διάστημα για την Ευρώπη του 2016 και η έκθεση της ΣΥΤΡΕ για μια διαστημική στρατηγική ε, δείχνουν πόσο μεγάλη σημασία αποδίδουμε. Λοιπόν, μιλήσατε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρετε τους τρέχον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε 12,2 δις για το Γαλιλαίο 7, για το Κοπέρνικο 4,7 και 1,3 για τη διαστημική έρευνα μέχρι το 2020. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι τοποθετήσεις Σα Ακούσαμε ότι θα, χρειαστεί ακόμη περισσότερο, θα χρειαστεί ακόμα περισσότερες επενδύσεις στο μέλλον η ανάπτυξη του, των δραστηριοτήτων μας στο διάστημα. Μιλήσατε για μερικές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ε, κομμάτια διαστημικών συντριμιών σε κυκλοφορία, ε, μιλήσατε για διαχείριση της, ε, της κυκλοφορίας στο διάστημα με ε, εκατοντάδες δορυφόρους που σχεδιάζεται να εκτοξευθούν στο διάστημα στο εγγύς μέλλον. Άρα έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε κατά τρόπο ικανοποιητικό την λειτουργία του διαστήματος. Δεν φτάνουν λοιπόν τα ε, ποσά που προβλέπονται για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με δεδομένη και την μείωση του συνόλου του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού κατά 12 δισεκατομμύρια ενώπιση του Brexit. Επομένως αυτό που θέλω να σας ρωτήσω εγώ είναι περισσότερα έξοδα θα έχουμε, θα χρειαστούμε άρα και περισσότερα δαπάνες να προβλέψουμε στους προϋπολογισμούς μας, στον προϋπολογισμό μας. Πρέπει να υπολογίσουμε την στάση των Αμερικανών ενδεχομένως ε, μπορεί να μας ε, κοστίσει κάτι η συνεργασία σχετική με την ανταλλαγή ε, πληροφοριών και δεδομένων με τους Αμερικανούς και επίσης η εμπορευματοποίηση του διαστήματος γιατί η Ευρώπη και διάφορα κράτη θέλουν να αναπτύξουν βεβαίως δραστηριότητες ως κρατικές οντότητες στο, διάστημα αλλά υπάρχουν και ιδιωτικές επιχείρησεις οι οποίες θέλουν να εκμεταλλευτούν εμπορικά το διάστημα. Ρωτώ λοιπόν υπάρχει μια στρατηγική στην Ευρώπη με βάση την οποία να υπάρχει η στόχευση της αντιμετώπισης, της διαχείρισης του ΣΥΠΗΝ αυτών των πρωτοβουλειών Φερρυπίν με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για το διάστημα. Ευχαριστούμε. Τώρα και η δική μου ερώτηση. Ακούσαμε πολλά για την ευρωπαϊκή αυτονομία, την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία ε, σε θέματα διαστημικής πολιτικής. Ε, Ακούσαμε και για τη θέση της Ευρώπης σε σχέση με τις είπα, το επίπεδο της συνεργασίας, ποια είναι η απαραίτητη συνεργασία επίσης και ο ανταγωνισμός σε κάποιο βαθμό στα θέματα αυτά. Αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για άλλες ε, συνεργασίες και εταιρικέ σχέσεις ε, και τάσεις που ακολουθούν αυτές τις συνεργασίες. Ποια είναι τα ωφέλη τους επίσης, ποιες είναι οι προκλήσεις και η ερώτηση μου, την ερώτηση μου την απευθύνω σε όλους τους ε, καλεσμένους μας. Θα ήθελα να μας απαντήσετε τώρα με τη σειρά που κάνετε τις παρουσιάσεις σας, οπότε πρώτος ο κύριος Αλάρετιε. Ευχαριστώ, θα μιλήσω γαλλικά. Λοιπόν, για την πρώτη ερώτηση, όσον αφορά τον πλήθος των δορυφόρων που απενεργοποιούνται και πόσα απόβλητα συνεπάγονται, το πρώτο ερώτημα είναι ότι ε, το πρότυπο ε, ISO 24113, ο σχετικός κανονισμός, ε, εισήχθη πρόσφατα. πολύ, δηλαδή δορυφόροι, χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τέλους και δεν είναι πλέον υπό έλεγχο. Πρέπει να τους ανακτήσουμε δηλαδή και γίνονται κάποιες πρωτοβουλίες σε ορισμένες περιπτώσεις ή δεν έχουμε καμία ε, στη ΣΥΠΑ δεν, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τίποτα. Στη ΣΥΠΑ ε, ένας Αμερικανός, Αμερικανικός δορυφόρος πέρυσι εξεράγει και δημιούργησε πολλά απόβλητα. Μετά έχουμε και τις δράσεις ε, χωρών όπως η Κίνα που χτύψαν με λέιζερ ε, παλιούς δορυφόρους πειραματικά για να δοκιμάσουν κάποια αμυντικά μέσα. Οπότε αυτούς που βρίσκονται σε τροχιά είτε τους ανακτούμε αλλά τα απόβλητα είναι στατιστικά στοιχεία. Υπάρχουν κάποια ε, μοντέλα που μας μπορούν να μας βοηθήσουν να προβλέψουμε πώς... ποιες είναι οι πιθανότητες σύγκρουσης με τα απόβλητα. Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ χαμηλής τροχιάς και γεωστατικής τροχιάς. Ε, υπάρχει κάποια πειθαρχία τώρα για τη γεωστατική, διότι θεωρείται σπάνιος εμπορικός πόρος, οπότε πολλοί δορυφόροι σήμερα τοποθετούνται σε τροχές στάθμευσης, ε, όπως λέγονται, που θεωρούν ότι έχουν υψηλή εμπορική αξία. Οι χαμηλέ τροχές είναι πιο δύσκολες. Οπότε το πρώτο είναι ότι πρέπει να υπάρχουν διεθνεί νομοθεσίε οι οποίε να εφαρμόζονται. Χρειάζεται δηλαδή ένα διεθνέ πλαίσιο ε, ενδεχομένω των ΗΠΑ και δεύτερον οι φορεί ε, όπω η UMATSAT δεν έχουν, που δεν έχουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν ε, για την απομάκρυνση από την τροχιά των παλιών του δορυφόρων να δράσουν εθελοντικά. Και τι έχουμε κάνει εμείς για τους δορυφορούς, τους παλιούς δορυφόρους με τόπο. Ε, θέλουμε να τους αποσύρουμε. Τα κόστη τώρα ανάκτηση των παλιών δορυφόρων ε, τώρα δοκιμάζονται, ε, κάνουμε τα πειράματα τεχνολογικά. Σε κάποιε ερωτήσει δεν θα απαντήσω γιατί δεν είμαι σε θέση να το πράξω δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Για το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος της EUMETSAT. Ε, για την εμπορευματοποίηση του διαστήματος, δεν μιλάμε για εμπόριο στο διάστημα, μιλάμε για το διάστημα ως εμπορικό χώρο. Για παράδειγμα, στη ΣΥΠΑ συζητάμε για την εμπορευματοποίηση διαστήματος της, ε, ενός κομματιού του διαστήματος και μάλιστα σήμερα οι βιομηχανοί προτιμούν να πληρώνουν υπηρεσίες ε, και να υλοποιούν την ανάπτυξή τους παρά να ε, βλέπουν να αναπτύσσονται υποδομές από το δημόσιο τομέα. Ε, το ίδιο συμβαίνει και στο... για τη Σελήνη. Αν ο κ. Τραμπ θελήσει να πάει στη Σελήνη, όπω ανακοινώθηκε πρόσφατα, μιλάμε για 20 ετήσεις επενδύσεις. Ε, αν η βιομηχανία λοιπόν πληρώνει υπηρεσίε για να αναπτυχθεί ε, υποδομή που χρησιμοποιεί η ίδια, αυτό είναι ενδιαφέρον οικονομικά. Αλλά υπάρχει κάποιο κίνδυνο γιατί οι Αμερικανοί πληρώνουν πολλά για να γίνεται με τέτοια ανάπτυξη μέσω τη αγορά υπηρεσιών, αλλά ξαφνικά μπορεί να βρεθούν με πολύ επιθετικές ε, ε, τιμολογίες στην αγορά. Αυτά ήθελα να πω. Ε, στα άλλα θα αφήσω να απαντήσουν οι συναδελφοί μου. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ο Διευθυντής Μπρουινέ από τη Γενική Διεύθυνση Grow. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις με τη σειρά που διατυπώθηκαν. Καταρχήν, ως προς την προβολή των προγραμμάτων. Όντω είναι μείζον ζήτημα το θέμα τη προβολή και της προώθηση επικοινωνιακά των προγραμμάτων. Θα πρέπει πρώτα όμως να δούμε ποιο είναι το κοινό στο οποίο μπορούμε να απευθύνουμε αυτή τη διαφήμιση στην προβολή. Για το Κοπέρνικος, για παράδειγμα, ενώ το σύστημα αρχικά θεσπίστηκε για να ικανοποιήσει θεσμικές, κυβερνητικές ε, δαπάνες, οι περιφερειακές θεσμικές, ε, λόγω της πολιτικής δεδομένων, αναπτύξαμε ένα οικονομικό οικοσύστημα, κυρίως γενικώς με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της εφαρμογής της πολιτικής των δεδομένων, της ανοιχτή πολιτικής ε, δεδομένων δωρεάν και γενικευμένης πολιτικής και δημιουργήσαμε κάποια μέσα, κάποια εργαλεία, ώστε ε, να, αξιο... φέρουμε την τέχνη, τη γνώση που υπήρχε και να την αξιοποιήσουμε. Γι' αυτό και ε, είχαμε πολλές διαστάσεις του Κοπέρνικους. Θα έχουμε και μία άλλη σειρά εξωτερικών δραστηριοτήτων που μπορεί να φαίνεται ανώδυνο ή ουδέτερο, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ε, κάποιες εξωτερικές δραστηριότητες, ε, όπως κάνουν οι Αμερικανοί, outreach activities, ε, το κάνουν και για την NASA οι Αμερικανοί. Θα κάνουμε και εμείς κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, στα πλαίσια του Κοπέρνικος θα οργανώσουμε διαγωνισμό για την καλύτερη φωτογραφία, τις καλύτερες φωτογραφίες από επιστημονική άποψη μπορεί να μην είναι ελκυστική μια τέτοια οργάνωση, αλλά από πολιτική άποψη και από άποψη εξοικείωση γνώση ε, του συστήματο και τη συμβολή του συστήματο, ε, μια τέτοια πρόσβαση είναι σημαντική. Γιατί κανεί ε, θα πρέπει για να κάνει τι φωτογραφίε του να έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Έτσι θα εξοικειωθεί με το σύστημα. Οπότε θα έχει ένα διαφημιστικό χαρακτήρα. Όπως γίνεται και με τους πολιτικούς προεκλογική τους εκστρατεία. Επίσης, έχουμε συνεργασία σε ό,τι αφορά το Brexit ε, του επιτελείου του κυρίου Μπαρνιέ και του επιτελείου το, της Βρετανικής κυβέρνησης, αλλά βλέπουμε ότι για το διάστημα δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση, καμία ειδική μεταχείριση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Θα δούμε πώς ε, θα αντιμετωπιστούν κάποια γενικά σημεία που αφορούν και το διάστημα και αν στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο διάστημα για να ρυθμίσουμε τη διακοπή της συνεργασίας ή τη συνέχιση της συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο στα υπάρχοντα προγράμματα. Τώρα, το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κυρία Καπέλα, δεν μπορώ εγώ να προεξοφλήσω μία μείζωνα πολιτική διαδικασία. Οπότε, ανάλογα με τους περιορισμούς που θα ισχύσουν και που τους απαριθμίσατε πολύ εύστοχα, θα πρέπει να γίνει μία ιεραρχική διαρρυθμίση. Μία ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και μια και υπάρχουν περιορισμού, θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα αν δεν ιεραρχήσουμε τι προτεραιότητες μα. Δεν είμαι εγώ όμως ο υπάλληλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολείται με την άμυνα και το διάστημα να κάνει αυτή την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Αν εσεί με ρωτήσετε, είναι σημαντική η άμυνα και το διάστημα, θα σα πω φυσικά ναι, αλλά δεν αρκεί να το πω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, όπω το είπατε και εσεί εμέσως και σα ευχαριστώ, Έχουμε κάποιους δορυφόρους ήδη σε τροχιά. Για τον Γαλιλαίο χρειάζεται κάποια ποσότητα για να λειτουργεί το σύστημα. Ε, και θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τους ανενεργούς φυσικά δορυφόρους και να έχουμε μια αλλεπάλλη χρήση δορυφόρων και αντικατάσταση. Στο πλαίσιο του Κοπέρνικους έχουμε έξι οικογένειες διαφορετικές δορυφόρων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δύο σε ε, τροχιά αυτή τη στιγμή. Οπότε το α και το β που είναι ήδη σε τροχιά θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία διαγωνισμού για τους επόμενους δύο δορυφόρους ε, γ και δ και θα πρέπει να εξασφαλιστεί κάποια αναλλαγή και κάποια συνέχεια. Οπότε, αν δημιουργήσουμε αυτό το νέο οικοσύστημα γύρω από τα δεδομένα του Κοπέρνικο και υπάρχει ένα οικονομικό κλάδο που θα αρχίσει να διαμορφώνεται, αυτό ο οικονομικό κλάδο εξαρτάται από τα δεδομένα που θα το δώσουμε. Εξαρτάται από τη δική μα τροφοδοσία με δεδομένα. Και αν κάποια στιγμή η ροή δεδομένων διακοπεί, θα θέσουμε σε κίνδυνο ολόκληρο το σύστημα που δημιουργήσαμε. Τώρα για τις εξαγωγές δεν νομίζω ότι υπάρχει, έχουμε σήμερα αυτό το πρόβλημα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος το θέμα των εξαγωγών. Και ως προς την ερώτηση της Προέδρου, επί του παρόντος, για το Γαλιλαίο έχουμε κάποιες συμφωνίες με την Ορβηγία και για το PRS έχουμε διαπραγματεύσει για συμφωνία με τις ΗΠΑ για ανταλλαγή δεδομένων. Στα πλαίσια του Κοπέρνικους μια ναι, και τα δεδομένα ήδη είναι ανοιχτά, προσιτά και ελεύθερα και δωρεάν. Διαπραγματευόμαστε με τρίτες χώρες. Έχουμε μέχρι στιγμή συμφωνία με την Αυστραλία και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά δρομολογούνται και άλλες 5-6 συμφωνίες. Οπότε έχουμε ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κόβων. Hub and Hub. δεν παίρνουν μέσω του διαδικτύου, αλλά είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των βάσεων δεδομένων μας. Οπότε διευκολύνουμε τη χρήση των δεδομένων, την πρόσβαση στα δεδομένα των Αυστραλών και των ε, Ινδονησίων, θα μας πείτε δωρεάν, ενώ φορολογούμενος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα χρηματοδότηση. Γιατί η απάντηση είναι απλούστατη. Με τα δεδομένα, χωρίς αλγόριθμο και χωρίς επεξεργασία, δεν πάτε πουθενά, δεν κάνετε τίποτα. Και αυτή τη στιγμή, δεδομένη τη ε, αρχαιότητα του Κοπέρνικου στην Ευρώπη, αυτό που κάνει του αλγόριθμου, στην επεξεργασία, και τη διαχείριση των δεδομένων οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και από τη στιγμή που συνάψαμε συμφωνία με την Αυστραλία, πέντε σημαντικοί πάροχοι Ευρωπαίοι άνοιξαν υποκαταστήματα στην Αυστραλία για την ε, επεξεργασία των δεδομένων. Οπότε εμείς έχουμε τις πρώτες ύλε και χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά κάποιος θα πρέπει να την μεταπεί αυτή την πρώτη ύλη και εκείνη η δική μας προστιθέμενη αξία και με τα δεδομένα Landsat όταν δεν δίνονταν δωρεάν, ε, έτσι λειτουργούσαν και οι Αμερικάνοι. Κύριε Γκάλερ, μιλήσατε για τις θεσμικές ανάγκες και τι εννοούμε, αν είναι στρατιωτικές ή πολιτικές, μη στρατιωτικές. Όντως προσπαθούμε να καλύψουμε όλο το φάσμα και της δυτής χρήσης και της στρατιωτικής χρήσης και της πολιτικής χρήσης. Για παράδειγμα, μερικές φορές έχουμε ε, εφαρμογές διτής χρήσης, ενώ αρχικά το σύστημα δεν είχε σχεδιαστεί για τέτοια χρήση. Για το Κοπέρνικους, για παράδειγμα, αν έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια, θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα στηρίζεται σε, δεδομένα υπέρυθρα θερμικά. σημαντικό ζήτημα για την ε, υγεία των φυτών, αλλά και για άλλους τομείς που αφορούν τη φύση. Τα ίδια δεδομένα, τα ίδια στοιχεία, με διαφορετική επεξεργασία, έχουν ενδιαφέρον ε, για στρατιωτική χρήση, για ασφάλεια. Γιατί με θερμικά υπέρθυρα δεδομένα μπορείτε να δείτε τον εχθρό που περνάει τη γραμμή σας, για παράδειγμα. Οπότε αρχικά μπορεί ο να είναι κανονικός, αλλά από την αλυσίδα επεξεργασίας δεδομένων μπορούμε να στραφούμε προς στρατητική ή προς πολιτική χρήση. Αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω και τον διευθυντή Dancing να δώσει τις απαντήσεις του. Ευχαριστώ πολύ και επιτρέψτε μου με τη σειρά των ε, ομιλητών να δώσω απαντήσεις για τον κύριο Στογεύσκη. Όντως είναι 4.500 οι δορυφόροι σε τροχιά και μόνο 1.500 ακόμα είναι λειτουργικοί. Οι 3.000 δηλαδή δορυφόροι είτε πια δεν λειτουργούν είτε είναι αλεξέλεγκτοι κιόλα. Σήμερα έχουμε κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για περιορισμό των διαστημικών αποβλήτων. Πρέπει να βγουν είτε κατά τρόπο ενεργό είτε παθητικό μέσα στα 25 χρόνια από την οτρανοποίησή τους ή δορυφόροι από την τροχιά. Ε, από αυτούς τους 1.500 ε, που σας ανέφερα οι περισσότεροι είναι από τις πρώτες μέρες του διαστήματος διαστημικής τεχνολογίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν για τον περιορισμό που έχουν αναπτυχθεί ε, θα πρέπει εν ώψη και των πολύ μεγάλων εκτοξεύσεων που προβλέπονται 600 μαζικά οι ε, να γίνουν πιο αυστηρές και μάλιστα υπάρχουν χώρες όπως αυτή η οποία σκοπεύει να κάνει την εκτόξευση των 600 ταυτόχρονα η οποία μας λέει ότι σκοπεύει να τηρήσει αυτούς τους κανόνες περί περιορισμού των ε, τώρα της 25 ετία δηλαδή περιορισμού των αποβλήτων. Εσείς κύριε Γκάλερ μιλήσατε για, το space, για, το, για αυτό το θέμα το οποίο και εμένα με ενδιαφέρει το Space ε, Situation Awareness, πολιτική στρατιωτική συνεργασία. Έχουμε στον Τάρνστατ εδώ και αρκετά χρόνια με τον Υπουργό Έρευνας Στόλτενμπερκ συγκεκριμένα έχει υπογραφεί η ιδρυτική πράξη και εγώ ε, σε αυτό αναφέρθηκα όταν είπα ότι έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας από τη δορυφορική τεχνολογία. Το 1967 ήταν 10 χρόνια μετά την εκτόξευση του ρωσικού, του πρώτου δορυφόρου, του Sputnik, ε, και δύο χρόνια μετά τους Αμερικανούς. 50 ε, χρόνια λοιπόν ιστορίας έχουμε. Δεν χρειάζεται να ξαναεφεύρουμε τον ε, τροχό. Τεχνογνωσία υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εσείς αναφερθήκατε στο Brexit. Κοιτάξτε, ο ΕΟΔ είναι διακυβερνητική οργάνωση. Έχουμε λοιπόν 28 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελβετία και η Νορβηγία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, που οι δύο πρώτες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. το Ηνωμένο Βασίλειο δεν, ε, δεν έχει φύγει ακόμα και έχουμε βέβαια και τον Καναδά και άλλα συνδεδεμένα μέλη. Στην τελευταία υπουργική διάσκεψη του Δεκεμβρίου του 2016 στη Λουκέρνη της Ελβετίας διαπίστωσα μεγαλύτερη προσήλωση στο έργο του ΕΟΔ από τον Ομένο Βασίλειο από ό,τι είχατε μέχρι τώρα δει. Και αυτό νομίζω θα αντικατοπτριστεί και στην οικονομική συμβολή του, συνδρομή του. Και πρέπει να επισημάνω στην Επιτροπή σας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό που συμβάλλει τα μάλα, 25% στο πρόγραμμά μας για την ευαισθητοποίηση του Awareness Program και ιδιαίτερα στην πρόγνωση την μετεωρολογική έχει του επίπεδου καταγραφή. Ε, ωστόσο, το διαστημικό υλικό μπορεί όχι μόνο να προκαλέσει ζημιές στην, ε, ε, εισερχόμενο στην ε, ατμόσφαιρα αλλά και στο διάστημα και αυτό το είδαμε στην σκοτίδα, σκοτία στο παρελθόν. Άρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ιδιαίτερου λόγους να ενδιαφέρεται για όλα αυτά. Η κυρία Κάπελ, μια και λείπει. Ας μιλήσω αγγλικά, θα μπορούσα να της γερμανικά μας ρωτάει πώς θα αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί στον προπολογισμό ε, χωρίς βεβαίως ε, να μπω στον ε, λεπτό πάγο της πολιτικής όπου εσείς είσαστε πολύ πιο αρμόδιοι θα απαντήσω το εξής ότι εξ όσων θυμούμε δαπάνες για το διάστημα έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλες χώρες που, έχουν την πρωτοπορία στο διάστημα ε, πολύ υψηλότερε από ότι οι δικές μας, αν μάλιστα συγκρίνουμε το μεικτό μας ΑΕΠ ή ε, αφιερούμενο ποσοστό ΑΕΠ στο διάστημα. Γιατί λοιπόν να μην είμαστε οι πρώτοι ως περιφέρεια. Γιατί να έχουμε λιγότερη ανάπτυξη των στρατιωτικών ή πολιτικών υποδομών μας προς όφελος των δικών μας πολιτών. Και επίσης σημειώνω ότι οι προσπάθειές μας έχουν να κάνουν και με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρήση των δυνατοτήτων. Μίλησε η κυρία Κάπελ για τους εκτοξευτές SpaceX των Ηνωμένων Πολιτειών και εμείς προσπαθούμε να είμαστε στο δυνατόν πιο αποτελεσματικοί ως προς τη δαπάνη και την επένδυση και ιδιαίτερα στον ΕΟΔΟ με τον κύριο Μπρουένερ, τον Γενικό Μετευθυντή, ο οποίος έχει αναπτύξει πλέον την ιδέα του διάστημα τέταρτη εκδοχή 4.0, ε, με προαγωγή και των ΣΔΙΤ της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα με μεγαλύτερη ευθύνη αλλά και βέβαια μεγαλύτερο όφελος από τη διαστημική δραστηριότητα κατά αναλογία προς όσα βλέπουμε να αναπτύσσονται στις ΗΠΑ Στην ερώτηση της Προέδρου τώρα. Εταιρικέ σχέσεις με άλλους και συνεργασία. Εγώ αυτό που θέλω να ζητήσω είναι το ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο να μας ε, υποστηρίξει ως προς την ανταλλαγή των δεδομένων γιατί αν δεν μπορέσουμε να μπούμε μέσα σε ένα σύστημα ανταγωνιστικό για την παρακολούθηση ιδιαιτέρως και καταγραφή των συντριμιών των αποβλήτων, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τις οικονομίες ε, που απασχολούν και την παρέμβαση βέβαια της κυρίας Κάπελ. Επομένως, συνεργασία που θα είναι προς το όφελος τόσο της ασφάλειας όσο και της οικονομίας. το μας βοηθήσει δηλαδή στο να εξοικονομήσουμε σημαντικούς πόρους, εάν μπορούμε να συνεργαστούμε σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βαν Όρντεν ήθελε να δευτερολογήσει. Ναι, ε, πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που αναχώρησα από την αίθουσα, αλλά χρειάστηκε να πάω σε μια άλλη συνάντηση πολύ γρήγορα. Ίσως να απαντήσετε ενώ δεν ήμουν εδώ. Δεν είναι ακόμα σε αυτά τα πράγματα για μένα. Ποια είναι η πρόβλεψη των δαπανών για το επόμενο ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο σε σχέση με την τωρινή κατάσταση. Μπορείτε να μας πείτε κάτι ή το απαντήσετε ήδη και δεν το άκουσα. Αλλά ήθελα να διευκρινίσουμε και ένα σημείο που ανέφερε ο κ. Ντένσινγκ ιδιότητα μέλους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ε, είναι κατά κράτος, ε, κατά, κατά, ε, κράτος όχι κατά μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και ίσως μόλις το επιβεβαιώσατε οπότε η σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος δεν αλλάζει με τον Brexit. Σωστά? Director Dancing, yes. And... Ο κύριος Ντένσινγκ και αξιότιμη κύριε πως θέλετε και εσείς να πείτε ναι να το επιβεβαιώσω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι τακτικό μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Τώρα, ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ε, επιφορτίζεται με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών, των ε, ενωσιακών διαστημικών προγραμμάτων. Έχουμε δηλαδή συμφωνίες για τον Καλλιό και τον Κοπέρνικους. Οπότε εκεί είναι λίγο γκρίζα η ζώνη. Κάπως θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να, δούμε πώς θα γίνεται αυτό όσον αφορά τις λεπτομέρειες. Αλλά όπως είπαμε το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξήσει τη συμμετοχή του στο ίσα σε σχέση με παλιότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το, τρία μέλη του πάνελ για το, πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους ε, σε αυτό το πρωινό κομμάτι της συνεδρίας της ΕΝΤΕ σε σχέση με τις διαστημικές πολιτικές και διαστημικές δυνατότητες και μέσα. Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν τους ε, προσκεκλημένους μας για να τους ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, just a few... Λοιπόν, λίγα λεπτά διάλειμμα για να αλλάξουν τα μέλη εδώ.